Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντα θα εστιάσουμε πραγματικά ε, στην Ευρωπαϊκή. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα στη συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει στις Βρυξέλλες σε 15 μέρες στην ε, Ολομέλεια. Η επόμενη εισήγηση μας ε, είναι η αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, η καλή μεταχείριση των ζώων ε, είναι κάτι το οποίο ε, αφορά όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την ευζοία των ζώων, αλλά οπωσδήποτε αφορά και τη δική μας ταυτότητα. Εμείς ε, πιστεύουμε ορισμένα πράγματα για τους εαυτούς μας, ορισμένα πράγματα για την Ευρώπη, για τον πολιτισμό μας, για το περιεχόμενο του πολιτισμού μας και η καλή διαβίωση των ζώων αντικατοπτρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Συνεπώς είναι πολύ βασικό να δείξουμε ότι εκτιμούμε ε, αυτό το σύνολο των αξιών. Τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας θέλησαν να αναθεωρήσουν το σχέδιο δράσης μεταξύ 2006 και 2010 κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής ε, με εισηγήτρια την ε, Μαρίτ Πάουλσεν αξιολογήθηκαν ορισμένα έργα και θέλω να πω ότι όταν εξέτασα όλες αυτές τις δράσεις ανάμεσα στο 2006 και 2010 και επίσης όταν είδα και το μέλλον δηλαδή από το 2011 μέχρι το 2015 κατανόησα ότι πρέπει να ενισχύσουμε ορισμένες υπάρχουσες νομοθεσίες σε αυτόν τον τομέα. Σήμερα Πρέπει να πούμε ότι ειδικά η οδηγία ε, για τους χείρους και για την ευζοία των χείρων ε, θέτει ορισμένα προβλήματα, προβλήματα αιώνια, τα οποία επανέρχονται συνεχώς. Το θέμα της μεταφοράς των ζώων, για παράδειγμα, πάντα επανέρχεται αυτό το θέμα. Ο έλεγχος των κανόνων, ο σεβασμός της νομοθεσίας και οι κυρώσεις ε, οι οποίες υπάρχουν ή θα έπρεπε να υπάρχουν. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά από τα όρια που θέτουν τα σημερινά ε, νομιοθετικά κείμενα. Θέλω να υπάρχει μια ε, θέαση σφαιρικότερη του προβλήματος για ε, ό,τι αφορά την προστασία των ζώων, κάτι το οποίο είναι μια από τις βασικές προδιαγραφές της Ευρώπης για την εσωτερική της αγορά με διάφορα επίπεδα τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά παντού. Πρόκειται για μια μεγάλη ανανέωση ουσιαστικά κάτι το οποίο θα ευνοούσε και τον ανταγωνισμό μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς δεν θα μπορούσε να έρθει σε ανταγωνισμό με τον γείτονά του βάσει του κριτηρίου της καλής διαβίωσης των ζώων. Θα πρέπει επίσης να δείξουμε εμείς ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλες απαιτήσει ε, σε αυτά τα θέματα. Χρειάζεται απαραίτητος μια προστασία για ό,τι αφορά τον αθέμητο ανταγωνισμό που προέρχεται από τρίτες χώρες στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων. Γιατί να έχουμε εμείς υψηλή στάθμη όταν έχουμε ε, έναν αθέμητο ανταγωνισμό από τις τρίτες χώρες ο οποίος δεν ελέγχεται. Ε, αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να πληρώσουμε όπως και πληρώνουμε για την προστασία των ζώων. Πρέπει να υπάρχει ένα όφελος. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης χρειάζεται ένα σύστημα, ένα δίκτυο για να εξηγιάνουμε το υπάρχον σύστημα με μια σωστή οργάνωση. Το θέμα είναι, ετέθη αυτό το θέμα, το αν πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα αρχή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συντονιστούν οι υπάρχουσες αρχές. Υπάρχουν πολλές επιστημονικές οργανώσεις οι οποίες εργάζονται ικανά αλλά δεν έχουν ικανό συντονισμό μεταξύ τους. Επίσης το θέμα των αντιβιωτικών, η χρησιμοποίηση των ε, αντιβιωτικών στην εκτροφή των ζώων. Δεν μιλώ μόνο για τους κινδύνους ε, που, θέτουν, που τίθενται από τα κατάλοιπα των αντιβιωτικών, αλλά πιστεύω ότι τα αντιβιωτικά είναι ένας γενικός κίνδυνος για όλους μας, διότι και για τα ζώα αλλά και για τους ανθρώπους είναι πρόβλημα τα αντιβιωτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέιβις, ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην νομοθεσία, σε ένα μέρος ε, νομοθεσίας που αφορά τις ε, ε, όρνηθες. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αναβαθμιστεί μέχρι του χρόνου. Σε πολλά εμπορικά κέντρα ε, αυτό έχει ένα πολύ ψηλό κόστος εκατομμυρίων. Οι γεωργοί έχουν επενδύσει έτσι ώστε η καλή διαβίωση των ζώων να αυξηθεί ως επίπεδο. Υπάρχει συμμόρφωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρξει μέχρι του χρόνου. Δεν νομίζω. Θα ήθελα να ρωτήσω τι θα κάνει η Επίτροπη έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση γιατί η συγγήτρια μιλά για απαγόρευση στην εμπορία ε, αυγών που δεν συμμορφώνονται με την ομοθεσία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν οι γεωργοί των κρατών μελών να διασφαλίσουν ε, την αύξηση αυτών των κανόν συμμόρφωσης και ίσων όρων πρόσβασης για όλους. Ο κύριος Ντάντουερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Πόλσεν για την έκθεσή της. Χαιρετίζω τη δουλειά που έγινε από τους διάφορους σκιώδεις εισηγητέ στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτού του θέματος, ε, ιδίως ε, της ομάδας μου και της συναδέλφου από την ομάδα μου. Υπάρχει διαφορετική ευαισθησία για αυτό το θέμα από χώρα σε χώρα. Όλοι οι παραγωγοί, οι καταναλωτές δεν έχουν την ίδια αντίληψη για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, Λίγο-λίγο η ευρωπαϊκή νομοθεσία καταλήγει στη δημιουργία ενός υψηλού προτύπου, το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα νομίζω στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και ιδίως για τον έλεγχο των εισαγόμενων προϊόντων. Αλλά όπως υπόθηκε ήδη, αυτοί οι κανόνες έχουν και ένα κόστος. Και κάθε μέρα αντιλαμβανόμαστε ότι το κόστος είναι ψηλότερο για τους καλλιεργητές, ε, για τους διάφορους εμπορευόμενους τη στιγμή όπου η κερδοφορία της γεωργίας ε, πλήττεται όλος ιδιαίτερος. Να μια δικαιολογία για την ΚΑΠ. Αν ξοδεύουμε κάθε χρόνο 100 ευρώ ανακάτοικο για να χρηματοδοτήσουμε την ΚΑΠ, τότε η ευημερία των ζώων ε, είναι σαν τους λόγους που δικαιολογούν αυτή την, αυτά τα έξοδα. Ο επόμενος ομιλητής παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Πόλσον ε, γιατί μας δίνει λύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι γεγονός ότι η υγεία των ζώων ε, προϋποθέτει την καλή διαβίωσή τους και τους καλούς βιολογικούς κανόνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαβιώσουν καλά στο φυσικό περιβάλλον και να μην αλλάζουν συνθήκες διαβίωσης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την ε, καλή διαβίωση των ζώων και συμβαδίζοντας ε, τα αιτήματα για την προστασία τους. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη την αναθεώρηση της τεχνογνωσίας για την εκτροφή των ζώων και την χρησιμοποίηση νέων αποδοτικών τεχνολογιών για την φυσιολογική ζωή των ζώων και για να μπορέσουν να είναι παραγωγικά μέσα στα πλαίσια της ασφαλούς διατροφικής αλυσίδας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα, α, τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις και κονδύλια έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε όλες, ε, όλες τις προϋποθέσεις για την καλή διαβίωση των ζώων και τα καινοτόμα στοιχεία και μέτρα. Θα πρέπει να βρούμε τις ε, βέλτιστες δυνατές ε, λύσεις για την κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε ένα πρόγραμμα σε αυτό το τομέα λαμβάνοντας υπόψη την καλή διαφύωση των ζώων σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχετε μόνο ένα λεπτό. κυρία Γερεμάκη. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι και, το επίπεδο διαβίωσης, αλλά και ε, το δικό μας επίπεδο ε, διαβίωσης ως Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής έλεγχος και υπάρχουν πολλά ε, ελλείμματα, ελληματικές πολιτικές. Μιλάμε για τη μεταφορά των ζώων. Ε, είδαμε ταινίες στην τηλεόραση που μας μιλάνε για μια ζωφερή πραγματικότητα και όλα αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με την καλή διαβίωση των ζώων. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει εντάχει να λάβει μέτρα έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει ε, την καλή διαβίωση και καλή μεταχείριση των ζώων. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, ευχαριστώ το Κοινοβουλίο και ιδιαίτερος την κυρία Πόλσον ε, για την πρωτοβουλία της να ετοιμάσει αυτή την έκθεση για την ευμερία των ζώων. Η έκθεση αυτή ε, αποτελεί ένα προβληματισμό για ό,τι έχει συμβεί, αλλά και έχει χρήσιμες ιδέες για τη μελλοντική μας στρατηγική για την ευημερία των ζώων. Το σχέδιο δράσης που υιοθετήθηκε το 2006 ήταν ε, βασικά μια επιτυχία. Διάφορες πρωτοβουλίες σωματοποιήθηκαν ε, για να δημιουργήσουμε μια σφαιρική ε, θεώρηση για την ευημερία των ζώων και η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής είναι γενικά ικανοποιητική. Η και η Κομισιόν ε, θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν όμως περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή της, προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του Chris Davis, θα απαντήσουμε γραπτός. Είναι δύσκολο να απαντήσουμε τώρα προφορικά. Αλλά εμείς είμαστε πραγματικά άγρυπνοι σε θέματα εφαρμογής σε θέματα δίκαιου ανταγωνισμού εξετάζουμε βεβαίως και τη σχετική νομολογία. Ε, μας ενδιαφέρει ε, ο σωστός ανταγωνισμός μεταξύ των Ευρωπαίων και μη Ευρωπαίων παραγωγών. Ε, η ευημερία των ζώων είναι ένα μη εμπορικό έλλειμμα, το μέλημα, συγγνώμη, το οποίο θα πρέπει μονίμως να προτάσουμε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Τώρα για το 2011-2015 θα υπάρξει ένα νέο σχέδιο δράσης. Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες ε, για την εκπόνησή του και η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα στρατηγική για την ευημερία των ζώων ε, μέσα στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης, λαμβάνοντας ε, υπόψη το κόστος για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, τις προσπάθειές τους για την ευμερία των ζώων. Όπως αναφέρεται, κυρία Πόλσον, στην έκθεσή σας, το σημείο, μάλλον το άρθρο 13 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ευημερία όλων των ζώων. Επίσης και την, ε, το δίκαιο για την ευημερία των ζώων όπου υπάρχει. Αυτό το δίκαιο θα μπορούσε να είναι το, η βάση για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες και τις νομοθετικές, αλλά και θα πρέπει να ενημερώνει και τους καταναλωτές ε, και θα πρέπει να κινητοποιεί και την ε, έρευνα υψηλού επίπεδου. Επίσης, ε, σας ευχαριστούμε για την ε, υποστήριξή σας για αυτά τα δίκτυα με την συμμετοχή των κρατών μελών και των stakeholders για να προωθηθούν οι πρωτοβουλίες για την ευμερία των ζώων. Συμφωνώ ότι η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να δει ε, το θέμα της ανταγωνιστικότητας, το κόστος και θα πρέπει να είναι συμβατή με τις υπόλοιπες πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη την βιωσιμότητα των προτάσεών μας ε, μέσα σε ένα σφαιρικό πλαίσιο. Η έκθεση λέει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι στο ύψος των φιλοδοξιών μας, ε, προβλέποντας επαρκείς πόρους για την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες